Συνάδελφοι, ήρθε η ώρα των ψηφοφοριών. Το πρώτο θέμα αφορά την έκθεση της κυρίας Ρέγνερ και την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Στίβ Μπριουά.